Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η ρύθμιση ανοίγει ένα νέο τρόπο για την ε, επίλυση αυτού του εθνικού ε, ζητήματος ε, στην Ευρώπη. Η προσπάθεια των μονομένων κρατών να επιλύσουν το θέμα των Ρωμά δεν έχουν οδηγήσει σε καμία επιτυχία. και αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πραγματικά κάτι το οποίο καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχετε το λόγο, κυρία Σίνκλερ. Είμαι κατά των διακρίσεων εναντίον ιουδήποτε ε, ε, τμήματος του πληθυσμού, αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω το ψήφισμα αυτό γιατί θέτει την ευθύνη καταπολέμησης των διακρίσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ενώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις εντελώς διαφορετικές καταστάσεις που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη μέσω μέτρων τα οποία θα πρέπει να λάβουν τα ίδια τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα αυτά τα οποία δεν συμμερίζονται τις αξίες μας ένας Ιταλός βουλευτής διώκεται γιατί πήρε μέρος σε παραστρατιωτικές ομάδες ε, εις βάρος των με παρανόμων μεταναστών. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν θα πρέπει να δημιουργείται σύγχυση λοιπόν και να μην πιστεύουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζονται οι μετανάστες το ίδιο επίπεδο υποστήριξης όπως αυτό στην Ιταλία. Van Heck. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι γεγονό ασφαλώς ότι όποιο αρνείται την αλήθεια και την ύπαρξη ενός προβλήματος δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Είναι γεγονό. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στο ψήφισμα αυτό για τους Ρωμά στην Ευρώπη Πρόκειται για ένα τελείω ανόητο έγγραφο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε οποιαδήποτε λύση. Δεν μπορούμε να προτείνουμε καμία λύση γιατί αρνούμαστε την ύπαρξη του προβλήματος. Θα πρέπει καταρχά να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν ε, τεράστια προβλήματα, μεγάλοι αριθμοί Ρωμά οι οποίοι κλείνονται έξω από την ε, κοινωνία μα και ότι αυτοί ευθύνονται για πολύ μεγάλο ποσοστό της μικρής και μεγάλης εγκληματικότητας. Η έλλειψη αξιών των κοινοτήτων Ρώμα αποτελούν τη ρίζα του κακού την, ε, για την, ε, το μη σεβασμό των αρχών που έχουμε. Ίσως να είναι μονομερή αυτά που λέω, αλλά θεωρώ ότι το ψήφισμα αυτό που ψηφίσαμε είναι μονομερές από την άλλη πλευρά και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν από μόνα τους πως αυτό το πολύ ρεαλιστικό πρόβλημα πρέπει να αντιμετώπιζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Σαμόρσκα. Señora Saborska, tiene la palabra. Señora Saborska. je m'excuse, Monsieur le Président. Ζητώ συγγνώμη, αλλά εγώ θέλω να μιλήσω για την έκθεση για την ανάπτυξη. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Όχι, λάθος σας έχουμε σημειώσει τότε. Κλάις. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την έκθεση αυτή, μία από πρόκειται για ένα ψήφισμα ακραίο, στο οποίο φαίνεται να έχει πατέντα το Κοινοβούλιο. Η κοινωνική στέρηση των Ρωμά αποτελεί αναφέρεται αποτέλεσμα του αποκλεισμού και των διακρίσεων. Αν επιβάλλουμε νέε ποσοστώσει, αν ανοίξουμε την κάνουλα με τα χρήματα, τα θα όλα. Η εμπειρία στην Ολλανδία έχει ωστόσο καταδείξει ότι ό,τι και να κάνουμε το μεγαλύτερο τμήμα της κοινότητας αυτής αρνείται να προσαρμοστεί και να ενσωματωθεί. Και ότι υπάρχει μεγάλη εκπροσώπηση στις στατιστικές για την εγκληματικότητα, αυτό οφείλεται στους ίδιους τους Ρωμά, όπου πολλές αξίες έρχονται σε αντίφαση με τις δικής μας και είμαι κατά οποιασδήποτε ευρωπαϊκής προσπάθειας να επιβληθεί στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση τέτοιων ατόμων από την επικράτειά τους και σε ό,τι αφορά την αντίσταση σε τέτοιες ε, εγκληματικές δράσεις. Ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε. Προσφέρετε του προπολογισμού 2011 δηλώσεις σχετικά με το κείμενο αυτό. Κύριε Μορκουνάη, το πρώτη. Σας ευχαριστώ υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό για μια σειρά λόγων. Αλλά κυρίως επειδή η απασχόληση μαστίζει ιδιαίτερα τους νέους, η σημερινή κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών απαιτεί να δοθεί έμφαση στην απασχόληση των νέων και θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε σε μια επένδυση στο μέλλον η τρέχουσα οικονομική κατάσταση υποδεικνύει ότι οι νέοι προτιμούν να ακολουθήσουν περαιτέρω εκπαίδευση παρά να αναζητήσουν ε, θέση απασχόλησης, ε, θέση εργασίας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε, να υποβάλουμε μέτρα και προτάσεις για τη σύνδεση της εκπαίδευσης αυτής με τις θέσεις εργασίας μετέπειτα. Για παράδειγμα, προγράμματα όπως το Εράσμους θεωρούμε ότι η προτεραιότητα αυτή θα πρέπει να μας καθορίσει και στην επόμενη νομοθετική περίοδο. Ο κύριος Φανέκε, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ και πάλι Πρόεδρε. Καταψήφισα την πρόταση αυτή. Καταρχάς γιατί διαφωνώ με τις προτεραιότητες που έχει προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση της μεταναστευτικής πολιτικής και ξέρετε τι εννοώ την οργάνωση τη ε, μεταναστευτική πολιτική όλων των κρατών μελών που τίθεται ως προτεραιότητα. Δεν συμφωνώ με αυτήν, αλλά καταψήφισα καταρχάς την έκθεση γιατί διασαφηνίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι υπέρ της πολύ απαραίτητης ε, γραφοκριτιοποίηση του συστήματος. Θα πρέπει να καταργήσουμε όλες τις υπηρεσίες οι οποίες είναι περιτές, ήταν περιτές ήδη στο παρελθόν. Και αντιθέτως το κοινοβούλιο αυτό ζητάει ακόμα πιο πολλές αποκεντρωμένες τέτοιες υπηρεσίες. Θεωρώ ότι έχουμε υπερβολικά πολλές και θα πρέπει να καταργηθούν κάποια από αυτά τα κάποιες αυτές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, το Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων. Ξέρετε πόσο στοιχίζουν όλα αυτά στον φορολογόμενο και τι νόημα έχουν, ποια πρακτική εφαρμογή έχουν. Ευχαριστούμε κύριε Φανέκε. η έκθεση για τι αντίρρες γραμμέ του προπολογισμού 2011 και ο Μποσινιόρε όσον αφορά την έκθεση και για τα άλλα τμήματα του προπολογισμού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με την ψήφο αυτή αποκτήσαμε ένα μέσο για την προστασία των καταναλωτών Διακόπτει ο κύριος Μονσινιώρε. Mm-hmm. Ναι, ναι, η έκθεση τρίπελ είναι. Όσον αφορά τις, τους προσανατολισμούς για το 2011 του προπολογισμού, τα άλλα τμήματα του προπολογισμού. Είχα ζητήσει να κάνω μια επεξήγηση ψήφου για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Ναι, είσαστε πάντα εγγεγραμμένος. Θα σας φωνάξουμε. Λοιπόν, ο κύριος Μπονσινιόρε πάλι. Ζούμε μια έκτακτη περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτή τη έκτακτη περίοδου πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Οι προπολογισμοί τα επόμενα χρόνια δεν θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο επεξεργασία όπω μέχρι τώρα. Η οικονομική κρίση δεν έχει τελειώσει ακόμα και δεν είναι κάτι που μπορούμε να αγνοήσουμε. Η πολιτική μου ομάδα και εγώ ίδιος υπερψηφίσαμε τους προσανατολισμούς για το προϋπολογισμό σήμερα, αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε τις πολιτικές ευθύνες στο μέλλον, να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις μεταρρύθμιση σε βάθος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα της δώσει τη δυνατότητα να επαναπροσανατολίσει την οικονομική της πολιτική, να διευρύνει την εσωτερική αγορά, να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις για την έρευνα, για την οικογένεια, Αλλιώς ο κίνδυνος θα είναι πάρα πολύ μεγάλος με εθνικές δράσεις συντηρητικές και χωρίς συντονισμό. Θα πρέπει να είμαστε πιο Ευρωπαίοι, λιγότερο εθνικιστές εφαρμόζοντα μια ουσιαστικά ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ κύριε Μπονσίνιορε. Άναν. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση σας ξαναβλέπω να προεδρεύετε κύριε Βιδαλκουάδρας. Ο Μαρκ Τουέν είπε ότι όταν το μόνο που έχεις είναι ένα σφυρί όλα γύρω σου αρχίζουν να φαίνονται σαν ένα καρφί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει, ξοδεύει όμως τα χρήματα των άλλων. Έτσι είχε πει και ο κύριος Φρίντμαν ότι είναι πολύ εύκολο να ξοδεύει τα χρήματα των άλλων. Και αυτό εξηγεί το τι συμβαίνει στην ε, Ευρώπη σήμερα. Όλα τα κράτη-μέλη θέλουν να προχωρήσουν σε δημοσιονομικές ε, μειώσεις. Προτείνεται στην ε, Ελλάδα μείωση του δημοσίου τομέα κατά 10% περίπου, 7% στην ε, Ιρλανδία και σε άλλες χώρες αντίστοιχα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται ασταμάτητα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δαπάνες, στη φορολογία και αυτό είναι απαράδεκτο σε αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα οι πραγματικά υπερβολικές δαπάνες μας οδήγησαν από τις κυβερνήσεις αλλά και από τα μεμονωμένα άτομα και τους οργανισμούς και τις εταιρείες κτλ. Λοιπόν, το ίδιο λάθος κάνουμε και εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο σήμερα. Σε ευχαριστούμε για αφορά την πολιτική για ποιοτικά γεωργικά προϊόντα και έχει το λόγο ο κ. Καλινόφσκι. señor kalinowski no. tiene la palabra el señor Mikolasik. O κύριος Μικολάσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα είναι κορυφαίας ποιότητας. Αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι είναι πιο ανταγωνιστικά στο παγκόσμιο προσκήνιο. Οι πολίτες της Ευρώπης και οι συνειδητοποιημένοι καταναλωτές θα πρέπει να διακρίνουν την ποιότητα αυτή. Γιατί δεν πληρούν μόνο τα πιο υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά και τις κτηνιατρικές ε, προδιαγραφές, αλλά σέβονται και τα θέματα της ε, ποικιλία και της ε, πολυμορφίας. Γι' αυτό είμαστε υπέρ των ευρωπαϊκών προϊόντων. Το λογότυπο αυτό θα αναγνωρίσει το έργο των Ευρωπαίων αγροτών και θα προστατεύσει τα προϊόντα αυτά στην παγκόσμια αγορά. Προκειμένου η Ένωση να μπορέσει να προσφέρει την ποιότητα αυτή, θα πρέπει να εξασφαλίσει τον εξυγχρονισμό των ε, εκμεταλλεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μορκουναϊτέ. Ψήφισα υπέρ του εγγράφου αυτού γιατί θεωρώ ότι η γεωργία με περιβαλλοντικά πρότυπα αποτελεί το μέλλον μας και θα πρέπει να την προωθήσουμε. Θα πρέπει να προωθήσουμε και τα περιβαλλοντικά αυτά φιλικά προϊόντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε ωστόσο να προάγουμε αυτού του είδους την γεωργική εκμετάλλευση, δεν θα πρέπει να ε, βιαστούμε σε ό,τι αφορά τους ε, γενετικά τροποποιημένους ε, οργανισμούς. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των περιβαλλοντικών προϊόντων αυτών και των γάμα τα όμικρων. Οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται στους καταναλωτές σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς αυτούς και θα πρέπει να μην κρύβεται τίποτα από τον καταναλωτή. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για όλους μας. Ευχαριστούμε. Ο κ. Αντωνιώτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σκοτά για την πολύ καλή του δουλειά. Νομίζω ότι η φροντίδα για την ποιότητα των γεωργικών μας προϊόντων αποτελεί προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋποθέτει επίσης την επιδίωξη και άλλων στόχων παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή την προστασία του καταναλωτή, την υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την προστασία της παραδοσιακής κληρονομιάς, την προστασία της υπαίθρου, και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων σε ε, διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό και υπερψηφίζω την έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ θετικό η έκθεση για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων να βασίζεται ε, σε πολιτικές επιδίωξεις της ποιότητας οι οποίες είναι πολύ γνωστές εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι και τα συστήματα προ... προέλευσης, εγγυήσεων δηλαδή σχετικά με την προέλευση των προϊόντων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε να χρησιμοποιούνται περισσότερο στο μέλλον και θα πρέπει να προσπαθήσουμε με ευκολότερους τρόπους να καταγράφουμε τα προϊόντα αυτά τα παραδοσιακά. Δεν βλέπω λοιπόν τον λόγο για τον οποίο το χρονοδιάγραμμα για την καταγραφή αυτών των προϊόντων να μην είναι ε, ο ίδιο, το ίδιο μάλλον το χρονοδιάγραμμα αυτό με το αντίστοιχο που χρειάζεται για τα προϊόντα με εγγυημένη γεωγραφική προέλευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να μην βομβαρδίζει αυτούς οι οποίοι ζητούν την καταγραφή των προϊόντων με άπειρες ερωτήσεις γραφειοκρατικές. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σκοτά για την προσπάθειά του. Να αναφερθώ στην τροπολογία 4 που ζητά τις ε, πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να παίρνει ο καταναλωτής. Και επίσης το θέμα της ε, υποχρεωτικής ετικετοθεσίας είναι και τα δύο αυτά επίπεδα μια σωστή επιδίωξη αλλά θα πρέπει να μην υπερβάλλουμε στην πληροφόρηση αυτή. Εμείς στην Βόρεια Ιρλανδία εξάγουμε προϊόντα στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η τροπολογία αυτή μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της Βόρειας Ιρλανδίας να αποστέλει προϊόντα σε συγκεκριμένες αγορές, στις οποίες σήμερα δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Δεν θα πρέπει να δημιουργούνται διακρίσεις λοιπόν εις βάρος ορισμένων κρατών μελών. Δημιουργεί πρόβλημα λοιπόν η τροπολογία 4, παρόλα αυτά η έκθεση είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να είναι ανοιχνεύσιμα, ασφαλή και υψηλή ποιότητα στα γεωργικά προϊόντα. signore. Ευχαριστώ. Με την έκθεση Σκότα έχουμε ένα επιπλέον μίσο για την προστασία του καταναλωτή. Είναι ένα στόχος τον οποίο αναζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα η προέλευση του προϊόντος θα πρέπει να γράφεται στα προϊόντα που προέρχονται από ε, κρέας, από γάλα και ε, από άλλα προϊόντα. και τα ζώα μπορεί να έχουν συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση μόνο εφόσον έχουν γεννηθεί, ανατραφεί και σφαγεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τη γεωργική παραγωγή. Αποδείξαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρά επί των προϊόντων με μοναδικό στόχο την εγγύηση της ποιότητας και της προσβασιμότητας στην ενημέρωση του καταναλωτή. Κάναμε σωστή δουλειά και συγχαίρω τους συναδέλφους οι οποίοι προσπάθησαν τόσο πολύ. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί της αρχής δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα σε ό,τι αφορά το λογότυπο ισότητα. Το βλέπουμε αυτό σε πάρα, ποιότητα. Το βλέπουμε αυτό σε πάρα πολλού τομεί. Αρκεί να μην χρησιμοποιούνται ω δικαιολογία για να μην σεβαζόμαστε τι επιλογέ των καταναλωτών. Δεν μιλάμε δηλαδή για τρόφιμα με περιορισμού ε, ω προ την ποιότητα, ω προ ε, το μέγεθο. Δεν θα πρέπει να τα πετάμε όλα αυτά όπω γίνεται συχνά στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα πρότυπα ποιότητα ω δικαιολογία για να απαγορεύουμε εισαγωγέ από τι τρίτε χώρε, από αναπτυσσόμενε χώρε. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή ε, τα λεφτά των προλογουμένων για ε, διεφθαρμένε ε, πολιτικές κυβερνήσεις. Θα πρέπει να εμπιστευόμαστε και τον καταναλωτή και της αγοράς, να εμπιστευόμαστε τον κόσμο. Και τώρα έχουμε τι επιπτώσει τη χρηματοοικονομική ε, κρίση για τι αντισώμενε χώρε. Δηλώσει σχετική. Έκθεση ο κ. Μικολάσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταψήφισα την έκθεση αυτή, γιατί όπως πολλές φορές ακούσαμε, η Ευρώπη στην έκθεση αυτή θέλει να επιβάλλει στον κόσμο, στις αναπτυσσόμενες χώρες, τη δική της αντιλήψη σε ό,τι αφορά την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία. Σύμφωνα με τον ορισμό της ΠΟΗ, μιλάμε για θέματα αμβλώσεων, λες και πρόκειται για θέματα οικογενειακού σχεδιασμού. Δεν μπόρεσα λοιπόν να υποστηρίξω την έκθεση αυτή. Αφετέρου πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν και κάποιες ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν εις όφελος των ε, αναπτυσσόμενων χωρών. Οι άνθρωποι αυτοί στις χώρες αυτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις ε, άσχημες αυτές ε, συνθήκες διαβίωσης των οποίων η ίδια ύπαρξη απειλείται πρέπει να παραδεχτούμε ότι παρά τις ε, προσπάθειες των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων δεν βοηθούνται γιατί εξακολουθούν να αυξάνονται τα ποσοστά νησιμότητας. Ευχαριστούμε κύριος ε, Φίλεξης. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της κρίσης στις φτωχές χώρες του κόσμου παρά το γεγονός ότι η έκθεση αυτή δεν αποτελεί, αν θέλετε, ριζοσπαστική λύση για τα προβλήματα των φτωχών χωρών, μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που περιλαμβάνει, γιατί τελικά είναι οι φτωχέ οι χώρε. Ε, ο φτωχό κόσμος είναι αυτό που υποφέρει και πλήττεται πιο πολύ από την οικονομική αυτή κρίση. Θα πρέπει να παρέχουμε κάθε μορφή αρρωγής που μπορούμε στις χώρες αυτές. Αλλά το εμπόριο, οι εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελούν επαρκή τρόπο υποστήριξης ε, των χωρών αυτών. Ουσιαστικά οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι αυτές που ωφελούνται πιο πολύ από κάθε άλλον από τις συμφωνίες αυτές. Οι μικροί καλλιεργητές, οι μικρές εκμεταλλεύσεις ε, υποφέρουν ακόμα πιο πολύ. Θα πρέπει λοιπόν παραπάνω πράγματα να κάνουμε για την υποστήριξη των χωρών αυτών. Η κυρία Ντότσου. Um, uh, uh, Καταψήφισα την παράγραφο 7 της έκθεσης αυτής και γιατί είδα ότι για μια ακόμη φορά το Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε μια τέτοια έκθεση έτσι ώστε έμεσα να υπογραμμίσει και να ενισχύσει το δικαίωμα στην άμβλωση και να προωθήσει την ατζέντα της αναπαραγωγικής υγείας εις βάρος της δημόσιας υγείας γενικότερα. Δεν είναι εδώ ο χώρος ο οποίος θα δείξει αν η πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι δυνατή ή όχι. Τα θέματα αυτά τα αποφασίζουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και η μεγάλη πλειοψηφία των Βόρειων Ιρλανδών θεωρούν ότι πρέπει να πιστεύουν στα δικαιώματα του του παιδιού. Ο κύριος Φανέκ, ευχαριστώ πρόεδρε και πάλι. Θα πρέπει ως κοινοβούλιο να σκεφτούμε όταν κάνουμε προτάσεις, ότι οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να είναι υπέρ πολιτικών που θα επιλύουν προβλήματα, όχι ε, λύσεων που θα διαιωνίζουν προβλήματα, γιατί υπάρχουν πολλές σοβαρές μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι η αυτόματη αναπτυξιακή βοήθεια πολύ συχνά οδηγεί σε επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, στην επιβράδυνση δηλαδή Τη ε, της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και όλα αυτά, ω Ευρωπαϊκή Κοινοβούλιο θεωρούμε δεδομένο αξίωμα ότι όσο πιο πολύ αναπτυξιακή βοήθεια δίνουμε στις ε, αφρικανικές χώρες, τόσο πιο πολύ τις βοηθούμε. Και μετά από δεκαετίες μαζικής ε, αναπτυξιακής βοήθειας, δεν έχουμε δει κανένα αποδεικτικό στοιχείο Αντιθέτως, πολλές αφρικανικές χώρες είναι σε πολύ πιο άσχημη κατάσταση σε σχέση με, τα, με την περίοδο μετά την απεικιοκρατία. Αυτό γιατί, γιατί πολλές φορές υπάρχει διαφυγή εγκεφάλων. Γιατί όμως ε, στην περίπτωση αυτή εξακολουθούμε να εμένουμε επί της μπλε κάρτας, η οποία θα επιθυμώσει περαιτέρω το πρόβλημα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σαμπόσκα. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν κατανοώ γιατί η αναπαραγωγική υγεία έχει τεθεί εκ νέου στην έκθεση αυτή για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης στις αναπτυσσόμενε χώρες και στην ανάπτυξη και συνεργασία. Το να υποστηρίξει κανείς την άμβλωση στα πλαίσια του οικογενειακού προγραμματισμού στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο το αποφασίζουν οι φορολογούμενοι. Και απ' την άλλη υπάρχουν φορολογούμενοι των οποίων τα χρήματα παρά τη θέλησή τους χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτούνται τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές. Οι αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να ζουν σε φτώχεια με συγκεκριμένη αποτυχία των προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού τα οποία έχει επιχορηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι στις σχέσεις μας με τις αναπτυσσόμενες χώρες βασική αρχή πρέπει να είναι η επικουρικότητα. Ο κύριος Χάνων εκ Κύριε Πρόεδρε, ήταν προβλέψιμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθούσε να επωφεληθεί από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα για να προωθήσει την ιδέα της εναρμόνισης των φορολογικών και οικονομικών πολιτικών. Είδαμε τις εκκλήσεις για πανευρωπαϊκούς φόρους, για ευρωπαϊκές επιτροπές, ο κύριος Βαν Ρόμπεϊ, οι επίτροποι, υπέρ της Ομοσπονδίας ε, συμφωνούν λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει νομισματική ένωση χωρίς οικονομική και πολιτική ένωση. Ο Κέινς έλεγε όποιος ελέγχει το νόμισμα ελέγχει και τη χώρα και είναι η μόνη στιγμή που συμφωνώ με τον Κέινς. Αλλά εν πάση περιπτώσει στην ουσία εδώ προβλέπεται στο κεφάλαιο 22 του α, Ευαγγελίου κατά, το, κατά Ματθαίο. Λοιπόν, και <clears throat> λέγει το Ευαγγέλιο ότι θα πρέπει ο καθένας ουσιαστικά να ασχολείται με αυτά τα οποία πρέπει να ασχολείται και όχι να προσπαθεί ε, να εισβάλλει σε άλλα πεδία και να παραβιάζει την ακαιρεότητα. Λοιπόν, τα του Κέσαρωστού και τα λοιπά και ο καθένας θα πρέπει να προσπαθήσει και εμείς δικαιωθήκαμε γιατί κρατήσαμε τη Στερλίνα. Ευχαριστώ. Γιατί πράγματι αγιοποιήσατε τις συζητήσεις κύριε Χάναν. Κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν βλέπει κανείς την έκθεση αυτή βλέπει πολλά κουρασμένα στοιχεία τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ στο παρελθόν σχετικά με την οικονομική κρίση. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, αλλά πολλές φορές ε, δεν βοηθάμε αυτούς που θέλουμε να βοηθήσουμε. γιατί μερικές φορές ε, όσο λιγότερα χρήματα τους δίνουμε τόσο λιγότερο βοηθάμε τις διαφθαρμένες κυβερνήσεις να παραμένουν στην εξουσία. Μου έλεγαν πέρυσι σε αφρικανικές χώρες που επισκέφθηκα ότι οι κυβερνήσεις αυτές ζουν μέσω της ευρωπαϊκής βοήθειας. Ζητάμε περισσότερες επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και όλοι συμφωνούν με αυτό. Παρ' όλα αυτά, εμείς προωθούμε νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες παρεμποδίζουν τις επενδύσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε τέτοιες χώρες. Και θέλουμε να βοηθήσουμε τους γεωργούς των χωρών αυτών, αλλά παρόλα αυτά σήμερα πήραμε αποφάσεις οι οποίες είναι υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης της κοινή αγροτικής πολιτικής που λειτουργεί αρνητικά για τις χώρες αυτές. Κάστλα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταψήφισα την έκθεση αυτή για δύο λόγους. Καταρχάς, με ενοχλεί το γεγονός ότι η Ευρώπη όλο και πιο πολύ, σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή πολιτική, ανοίγει τις κάνολες και όλο και πιο πολλά ψηφίσματα και εκθέσεις ε, εκδίδει κατά δεύτερον ψήφισα κατά γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άσχημο το γεγονός ότι προσπαθούμε να κάνουμε υπεριαλισμό πολιτισμικό στα κράτη της δεύτερου και τρίτου κόσμου πώς πρέπει να κάνουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε την άμβλωση ως μέσο και λυπάμαι που το τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, τάσσεται υπέρ της, των αμβλώσεων με αυτόν τον πολύ όμορφο όρο της αναπαραγωγικής υγείας, το οποίο δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι πρόκειται για φόνο ουσιαστικά των αγέννητων παιδιών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να αποφεύγονται τέτοιοι όμορφοι όροι οι οποίοι ουσιαστικά είναι υπεριαλιστικοί. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βίβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι ανόητη η έκθεση αυτή. Είναι άσχετη η έκθεση αυτή. Υποτίθεται ότι προσπαθεί να καλύψει όλες τις καταστάσεις που δημιουργούνται στον κόσμο σε όλες τις ε, όλα τα χρηματοπιστωτικά κέντρα και τα χρηματιστήρια. υπάρχουν στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, πάρα πολλά, ε, πάρα πολλά στοιχεία πλούτου, τα ακίνητα σαν παράδειγμα, τα οποία δεν είναι πουθενά εγγεγραμμένα, είναι εκτός της νομικής δομής των χωρών αυτών. Υπάρχουν εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις που δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένες. Και αν θέλει κανείς να μάθει πόσα χρήματα παράγει ο αναπτυσσόμενος χώρος, θα μπορούσαμε να μιλάμε για 800 δις κεφάλαια. Γιατί να μην κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να παραμένουν στις ε, υποανάπτυξης χώρες. Θα πρέπει ίσως κατά τον εισηγητή να εισάγουμε το φόρο τόμπινγκ και να τους κάνουμε τη ζωή πιο δύσκολη και να δώσουμε χρήματα από την άλλη σε ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να τα κλέψουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δεν θα ήθελα να συμπεριληφθεί παράγραφος 7 στο κείμενο. Είχαμε ψήφο κατά στην πολιτική μας ομάδα, αλλά η προσωπή μας τελικά κατεψήφισε γιατί τα περί δικαιωμάτων αναπαραγωγικής υγείας είναι συνώνυμα της άμβλωσης. Επομένως, όπως και άλλοι, που έλαβαν ε, το λόγο. Είμαι και εγώ κατά αυτή τη διάταξη. Ευχαριστούμε κύριε Κυρλή, ο Πρόεδρο. Και τώρα, δηλώσει για την εκθέση Σικλούνο. Κύριο Μέσο Σμιτ. Er Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο Βανικό Κόμμα ψήφισε κατά της έκθεσης αυτής και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια σειρά σκέψεων που αναφέρονται, για παράδειγμα στο 27, στο σημείο 27, όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να οδηγήσουμε, να οδηγήσουν τα μέτρα αυτά υπέρ της σύγκλησης στις πολιτικές αυτές. Αλλά χαίρομαι που υπάρχει τουλάχιστον ε, ειλικρίνεια εκ μέρους του εισηγητή. Το ευρώ δημιουργήθηκε για να δοθούν πιο πολλές πολιτικές ε, κατευθύνσεις σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Σε όλους τους οικονομικούς τομείς θα πρέπει να υπάρξει εξίσωση ουσιαστικά. Και λένε τώρα οι οικονομολόγοι στη Φραγκφούρτη στους Έλληνες τι θα πρέπει να κάνουν σε ό,τι αφορά την πολιτική τους, την οικονομική της πολιτική. Και θα ακολουθήσουν Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και το καθεξής. Και είναι σαφές λοιπόν γιατί η Δανία θέλει να παραμείνει εκτός της Ευρωζώνης. Θέλουμε να ασκούμε τη δική μας οικονομική πολιτική. Δεν είναι θέμα άλλων εθνικότητων αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. 7 Απριλίου, τη Δετάρτη, στη 2.30 επαναλαμβάνεται η Σύνοδος, η δική Σύνοδος για την εξέταση των αποτελεσμάτων